Κολλήγινο, κολλήγιν. Τα Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Selbst der Auswärtige Ausschuss verdient sich im weiten Rund des Plenarsaals, aber das soll uns nicht daran hindern. Χρησιμοποιούμε την τεράστια αυτή αίθουσα, αλλά αυτό βεβαίω δεν πρέπει να μα εμποδίσει. Διαπιστώνω πω δεν υπάρχουν αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Διαπιστώνω επίσης πως εδώ πέρα μόνο προσφέρει το χώρος για γενεθλίων και άρα ε, βαρώνει άστον. Χαίρομαι για το ότι αφιερώνεται χρόνο ενώ στη χώρα σας ε, θα πίνατε τσάι τέτοια ώρα γιατί βεβαίως σήμερα είναι τα γενέθλια της ε, Λέδης Άστον να τα εκατοστήσετε. Äh, Τώρα περνάμε στην ε, τακτική ανταλλαγή απόψεων με την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Σήμερα ειδικά ασχολούμαστε με τα ζητήματα της διάσκεψης Γκίμνιχ στην Κόπενχάγη και τα ζητήματα του Συμβουλίου που θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε βέβαια και ζητήματα Μέσης Ανατολής, Συρία, συνεργασίας με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Ιεμένη, Ευρωπαϊκή Ένωση Ασία, τις σχέσεις αυτές και την Συμφωνία Συνεργασίας και Σύνδεσης αλλά και Φιλίας αλλά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με το νέο μέσο Εταιρική σχέσης ένα τομέα που θεωρώ πως είναι ένα νέο σημαντικό πολιτικό μέσο εξωτερικής πολιτικής στην διάθεση της ΥΠΑ της εκπροσώπου και βεβαίως ε, το οποίο θα διαμορφώσουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο. Τα θέματα είναι πολλά και σημαντικά και έχουμε και τη Λευκορωσία και τις, κυρώσει, τις κυρώσεις, τη Συρία και ίσως το πιο επικίνδυνο τα ζητήματα δηλαδή ε, που σχετίζονται με το Ιράν και το πυρηνικό ζήτημα και με ποιο τρόπο μπορεί να αποφευχθεί μια μεγάλη κρίση εάν οι 5 συν 1 και εδώ πέρα θεωρώ πως παίζει σημαντικό ρόλο η κυρία Άστον ε, είναι σε θέση όχι μόνο να ε, διαπραγματευτούν αλλά να καταλήξουν και κάπου αλλά αυτό νομίζω πως ε, βεβαίως επαφίεται και στην άλλη πλευρά. Σημειώνω πως σε αυτή την κρίσιμη φάση είστε διαθέσιμοι να μας παρουσιάσετε την ε, θέση σας. Έχετε λοιπόν το λόγο. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας σας πάρα πολύ για τις ευχές σας για τα γενέθλιά μου δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ μαζί σα. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω λέγοντα κάτι σημαντικότατο για μένα, διότι θλίβομαι από την στρέβλωση των χθεσινών μου σχολείων στην εκδήλωση. Ε, κύριε Πρόεδρε, καταδικάζω ανεπιφύλακτα τις φοβερές δολοφονίες στο σχολείο Ζεχατόρη στην ε, Τουλούζη και απευθύνω συναισθήματα συμπαθίας προς τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων προς το λαό της Γαλλίας και την εβραϊκή κοινότητα. Χθες δεν έκανα κανένα παραλληλισμό μεταξύ αυτής της τραγωδίας και γεγονότων αλλού στη Μέση Ανατολή. Ε, κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε διάφορα θέματα προς συζήτηση σήμερα και αν επιτρέπετε στα αρχικά μου σχόλια θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω μια εικόνα ε, που αφορά αυτά τα γεγονότα και να σας δώσω μια γεύση, αλλά σίγουρα στην συζήτησή μας, όπως πάντα, θα μπορέσουμε να μπούμε σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσω με το Γκίμνικ στην Κοπενχάγη, διότι κάποια από τα θέματα που θίξατε σωστά, Πρόεδρε, ε, συζητήθηκαν. Ε, εξετάσαμε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας ήταν πώς η εξωτερική μας πολιτική θα ασκηθεί στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς θα επιφέρουμε αλλαγές σε τρίτες χώρες μέσω πιέσεων και κινήτρων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εν συντομία να σχολιάσω κάθε θέμα. Όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική, στο παρόν κλίμα πρέπει να ακολουθήσουμε στρατηγική προσέγγιση και να χρησιμοποιήσουμε και τους πόρους που γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν τον καλύτερο τρόπο όταν αποδίδουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή διάφορα ζητήματα στα οποία είμαστε ισχυρότεροι ως 27. Επιβεβαιώνω τις προτεραιότητες που είχα καθορίσει στις αρχές που είχα αναλάβει τη θέση αυτή, ότι θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εξωτερικής πολιτικής, να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά την πολιτική γειτονία, εκεί θα κρυθούμε και να αναπτύξουμε εταιρικές σχέσεις με τους ε, διάφορες χώρες για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Ε, συνεργασία, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας αποτελεσματικότερα. Επί παραδείγματι, η κοινή εργασία μεταξύ των ε, ΤΣΕΟΚ και των κατών μελών όσον αφορά το Νότιο ε, Σουδάν και να δούμε πώς μπορούν οι αντιπροσωπείες να βελτιώσουν τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη και να δώσουμε και χώρο στους εθνικούς ε, διπλωμάτες αντιπροσωπείες να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς ε, οίκους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις εθνικές αντιπροσωπείες ώστε εκεί να μπορούν να συναθρίζονται και να επιτυχάνουμε οικονομία κλίμακας και καλύτερα αποτελέσματα μέσω συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, όπω προανέφερα, συζητήσαμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ συχνά το έχω περιγράψει σαν ένα ε, νήμα, μύτο τη Αριάδνη που διατρέχει όλε μα τι δράσει. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω στην Επιτροπή του προτιθέμεθα να προτείνουμε ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν ένα τμήμα του πακέτου για να εφαρμόσουμε αυτά που αναφέρει η κοινή ε, δήλωση. Θέλουμε να έχουμε σχέδιο δράση. Θέλουμε να έχουμε προσανατολισμό όσον αφορά τη δράση που ακολουθούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε και πολιτική δήλωση σχετικά με τα προσεπίτευξη ε, έργα που θέλουμε να κάνουμε και θα θέλουμε στενή συνεργασία μαζί σα, Ό,τι κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα όσων κάνουμε. Δεν θα πρέπει να είναι κάτι που εφαρμόζουμε μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτή η πτυχή στα πάντα. Συζητήσαμε την ε, ανεξιθρησκεία, ε, την ελευθερία του να πιστεύει κανείς ότι θέλει, περιπλοκότατο θέμα, αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές μειονότητες και αναγνωρίσαμε τη σημασία της συνεργασίας μαζί τους, αλλά στα πλαίσια αντιμετώπισης κάθε μορφής διάκρισης κατ' εκείνων που έχουν κάποια πίστη και εκείνων που δεν, έχουν, δεν πιστεύουν σε κάτι. Συζητήσαμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο σύνολο που υπάρχει μεταξύ μόνος από τη μια πλευρά ε, και συνεργασίε και προσπάθειε από την άλλη. Πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσει με κάποιε χώρε για να υποστηρίξουμε του στόχου που θέλουμε να πετύχουμε. Και να υποστηρίξουμε όμω τι αξίε, τι απόψει και τι πεπιθήσει μα. Έχουμε ένα φάσμα διαφόρων μέσων στη διάθεσή μα από μέτρα περιοριστικά που πιστεύω ότι άλλαξαν τη Μπούρμα και το Μιανμάρ ε, θα μπορούμε όπως κάναμε να ανακαλέσουμε τους πεζοσφαίρους από τη Λευκορωσία. Αυτά είναι τα αρνητικά μετά μπορούμε να δώσουμε θετικά κίνητρα στην πολιτική γειτονία. Ε, το λέμε for more for more. Δίνουν περισσότερα για να κερδίσουν περισσότερα. Οι κυρώσει προσελκύουν την προσοχή των μέσων ενημέρωση, αλλά ποτέ δεν διαχωρίζονται από τι ευρύτερε πολιτικέ πρωτοβουλίε. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε τι συνέπειε των κυρώσεων από άλλε πρωτοβουλίε που μπορούν να ασκήσουν επιρροή επί ενό καθεστώτο ή μια καταστάσεω. Οι κυρώσει δεν εφαρμόζονται ποτέ μεμονωμένα και δεν θα πρέπει να κρίνονται απομονωμένα. Ε, σύμφωνα και με την έκθεση του Sir Graham Watson όσον αφορά τι κυρώσει εκ μέρου του ε, Κοινοβουλίου. Εκεί αναφέρονται παρόμοια. Ε, όσον αφορά τα κίνητρα έχουμε πολλά. Έχουμε την προσέγγιση περισσότερα για περισσότερα. Έχουμε και τα τρία μη, χρήματα, κινητικότητα, πρόσβαση στην αγορά, στα αγγλικά τρία μη. Και θέλουμε να υπάρχει συνεργασία στο εμπόριο και θέλουμε να συνεχίζεται και ο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών ή με την αντιπολίτευση στι διαφορέ χώρε, Αυτό ισχύει στη Λευκορωσία και ισχύει και στη Συρία και αναπτύξαμε μια νέα έννοια, νέες έννοιες της ομάδας κρούσης. Το χρησιμοποίησαμε στην Τινησία και στην Ιορδανία. Θέλουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο να έχουμε του οικονομικούς φορείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα είναι μαζί με εκείνους που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη οικονομική και πολιτική για να βοηθήσουμε τις χώρες που περνάνε περίοδο αλλαγής και μεταβαίνουν από μια μορφή διακυβέρνηση σε άλλη. Και όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε θέλουμε να συζητήσουμε τα θέματα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, Συνθήκη της Αβώνας, έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διάφορα μέσα για την εφαρμογή πιο συνεπούς ε, πολιτικής. Και έχουμε τεράστιες δυνατότητες εκεί μέσω των ε, διαφόρων μεθόδων που διατίθεται. Αλλά η αξιοπιστία μας εξαρτάται από τα επαρκή εργαλεία για να εφαρμοστούν οι προτεραιότητες. Αυτό τι σημαίνει και θα πρέπει να συμπεριλάβω και τους στόχους χιλιετίας αυτό, τους αναπτυξιακούς, και στα πλαίσια τη πρότασή μα θα εξακολουθούμε να είμαστε μεγαλύτεροι υποστηρικτέ στον κόσμο των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων μέσων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη και του Μέσου για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Θέλουμε επίση να είμαστε και εταίροι που διαλέγουν οι γειτονέ μα στην πολιτική γειτονία. σε ανταπόκρισή μα στα γεγονότα, στα πλαίσια τη ε, Αραβική Άνοιξη ε, έδειξε τι προστιθέμενη αξία που να προσφέρουμε και αυτά θα υποστηριχθούν από σωστά χρηματοδοτούμενα μέσα για την πολιτική γειτονή της Ευρωπαϊκής Έχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο διάφορε προκλήσεις, η αλλαγή του κλίματο, η μείωση τη φτώχεια, ο αφοπλισμό και πολλά άλλα θέματα. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με στενή συνεργασία με χώρε του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να προωθεί τα συμφέροντά τη όλο τον κόσμο και να εμβαθύνει τη συνεργασία τη με του εταίρου τη το μέσο για την δυτική σχέση είναι μια σημαντική καινοτομία του πακέτου και είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι σίγουρο. Η Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε έχει κεντρικό ρόλο να παίξει στις διαπραγματεύσεις ε, για αυτό το θέμα και τη συνέχεια θα δοθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες της Ένωσης ότι είμαστε υπεύθυνοι, ότι είμαστε ελεγχόμενοι όσον αφορά ε, τα χρήματα που ζητούμε για τα επόμενα χρόνια. Για τον προπολογισμό θα πρέπει να πετύχουμε πράγματα για τα χρήματα που θα θέτουμε μέσω θέση προτεραιοτήτων. Εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ε, ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κοινή φιλοδοξία με εμά να έχουμε πιο ε, επιφανή ρόλο όσον αφορά το παγκόσμιο προσκήνιο και ελπίζω ότι μπορώ να προσβλέπω στη δική σα υποστήριξη όσον αφορά το πολιετέ αυτό πλαίσιο. Πολύ σύντομα θα ήθελα να μιλήσω για τις σχέσεις που έχουμε με τις περιφερειακές οργανώσεις. Και αυτό ισχύει με τον αραβικό κόσμο, ιδίως στην παρούσα περίοδο. Ξέρουμε ότι οι περιφερειακές λύσεις απαιτούνται προκειμένου να επιληθούν περιφερειακά προβλήματα. Έχουμε συνεργαστεί με την Ένωση για τη Μεσόγειο που δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αποτελεί μοναδικό φόρουμ όπου συμμετέχουν 43 εταίροι και από κοινού θέτουν κοινέ στρατηγικές μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η απόφαση να ληφθούν αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταφέρει να μας κάνει να είμαστε πολύ πιο συνεπείς ε, στη δράση την οποία έχουμε. Και η Ευρωμεσογειακή ε, Συνέλευση καταφέρει επίσης να έχει μια πολύ σημαντικότερη προοπτική όσον αφορά και τις δύο όχθες της Μεσογείου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχει κάνει και θα κάνει στη διαδικασία αυτή. Και ξέρω ότι με τη συζητήση του κυρίου Σούλτ που είχαμε με τον κύριο Σούλτ ότι και αυτό έχει δεσμευτεί εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία όσον αφορά το ζήτημα της Λιβύης, τη συνεργασία που έχουμε με την ομάδα του Καΐρου και θέλουμε την, να πετύχουμε τη συνεργασία της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αραβικού Συνδέσμου και μέσω της εργασίας που κάνουμε με τους εταίρους αυτούς έχουμε πλέον μια ομάδα η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της Συρίας. Επίσης έχουμε δώσει ε, συγκεκριμένη υποστήριξη, όπως ξέρετε, βοηθώντας τον Αραβικό Σύνδεσμο να δημιουργήσει την δική, της, τον δικό, την δική του ομάδα υποστήριξης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα αυτή και ο οποίος βοηθήσει να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ε, η συνεργασία που έχουμε με την ομάδα των χωρών του κόλπου είναι πάρα πολύ καλή, ιδίως όσον αφορά την Ιεμένη. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις ανάμεσα σε μένα και στον Γενικό Γραμματέα και για αυτό το ζήτημα και για άλλα ζητήματα. Ξέρετε, το Συμβούλιο Συνεργασίας για τις χώρες του κόλπου θέλει να δημιουργήσει πιο σημαντικούς δεσμούς για τα κράτη-μέλη που τα απαρτίζουν και ακολουθούν ένα μοντέλο ολοκλήρωση το οποίο μοιάζει με αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται λοιπόν τη δική μα συμπερογνωμοσύνη προκειμένου να πετύχουν το στόχο αυτό. Αναφέρθηκα επίσης στον Οργανισμό της Ισλαμικής Συνεργασίας για την εργασία που γίνεται για τη Συρία, μια ομάδα επαφή που έχουμε δημιουργήσει. Η πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα στην Συρία στις 23 Φεβρουαρίου και ε, έχουν γίνει και άλλες επαφές έκτοτε. Οι αλλαγέ τώρα στο Μαγκρέμπ, οι επικείμενε αλλαγέ στην Αλγερία δημιουργούν τι απαραίτητε συνθήκε για ενωμένη συνεργασία για τι χώρε του Μαγκρέμπ και η συμμετοχή μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση στις, στην συνεδρίαση 5 συν 5 δείχνει επίση την δική μα ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά ζητήματα τα οποία θίξατε κι εσεί στην αρχή του λόγου σα, κύριε Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό και το πιο επίγον είναι η Συρία. Προτεραιότητά μας, όπως το γνωρίζετε, είναι να σταματήσει η βία και να υπάρχει πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς κανένα εμπόδιο. Και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία, την Κίνα, με τους αδέλφους μας στο Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί η απαραίτητη οδός ανθρωπιστική βοήθεια και θα πρέπει να πετύχουμε μια ικανοποιητική λύση. Στις 24 Φεβρουαρίου συνεδρι... Ε, συν... μετήχα σε συνεδρίαση με την ομάδα των φίλων της Συρίας και σε προηγούμενη συνεδρίαση που είχε γίνει επίσης στο Λονδίνο. Και στις δύο επαφές υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνένεση προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο καθεστώς στη Συρία. Και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την πίεση αυτή και στις επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε στο μέλλον. Με τη συνεργασία του πρώην Γενικού Γραμματέα Κόφι Ανάν και στις ε, τηλεφωνικές επαφές που είχα μαζί του, υποστηρίζω στικά τις προσπάθειες που κάνει, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, να σταματήσει η βία και προκειμένου να καταφέρουμε να, προωθή, να προωθήσουμε μια πολιτική λύση. Χαιρετίζω την έκβαση της Υπουργική ε, Συνεδρίασης ε, του Αραβικού Συνδέσμου και τη συμφωνία στην οποία έχουν καταλέξει με τον Υπουργό Σαγγελά για τα πέντε αυτά συγκεκριμένα σημεία τα οποία συνάδουν και με τη δική μας την πολιτική. Προφανώς θέλουμε και επιπλέον μέτρα, επιπλέον κυρώσεις και άλλες δυνατότητες. Συνεχίζουμε την πολιτική μας κατά του καθεστώτος και όχι κατά των πολιτών και συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας με την Συριακή Αντιπολίτευση όπου λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμός των δημοκρατικών αρχών σε όλες τις επαφές που έχουν με τις ομάδες αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες της Συρίας ότι μέσω της Ένωσης θα καταφέρουμε να βρούμε μία λύση. Υπάρχουν ε, τρία κράτη-μέλη που έχουν ε, φύγει από την χώρα, που έχουν ε, σταματήσει δηλαδή, τις διπλωματικές επαφές και δύο οι οποίες θα το κάνουν στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε πάντως να διατηρήσουμε τις επαφές μας και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς στην κατάσταση. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκαμε και στην κατάσταση όσον αφορά το Ιράν και το πυρηνικό ζήτημα της χώρας αυτής. Γνωρίζετε ότι έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί μία λύση στα πλαίσια του E3 plus 3 και στα πλαίσια της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις 6 ε, Μαρτίου συζητήσαμε τον κύριο Τζαλίλη και νομίζω ότι απεστάλλει αμέσω η επιστολή σε εσά, κύριε Πρόεδρε, και εμεί επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μα για συνομιλίε, γνωρίζοντα όμω ότι θα πρέπει να απαντήσει και το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα και θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, προτού γίνει οτιδήποτε άλλο. Οι προσπάθειέ μα προκειμένου να επιστρέψει το Ιράν στο τραπέζι των πραγματεύσεων ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικέ Έχουμε συνεργαστεί και με την ε, διεθνή κοινότητα για να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχουμε έντονη συνεργασία με όλους του συναδέλφου μας και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τρίτες χώρε σε όσους έχουν συγκεκριμένο συμφέρον ε, για να εμπλακούν στις ε, κυρώσεις που έχουμε επιβάλει. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτές οι κυρώσεις. Επίσης αναγνωρίζουμε βεβαίως πως οι πρόσφατες συζητήσεις με το Ιράν μας φέρνουν τώρα σε ένα σημείο στο οποίο είμαστε φιλόδοξοι και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να τις επαναλάβουμε. Και θα έχετε δει πως ε, σήμερα φιλεξένησα τους πολιτικούς διευθυντές των ε3 συν 3 για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τις ε, δυνατότητες διαπραγμάτευσης στο μέλλον. Ξέρω επίσης πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αναγνωρίσει το πόσο τρομακτική είναι η κατάσταση ανθρωπιστική στο Ιράν. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ε, δηλώσεις ε, και ζητάμε να σταματήσει η να υπάρξει ένα μορατόριο όσον αφορά την θανατική ποινή, όχι μόνο στην περίπτωση της κυρίας Ανστιάνη, αλλά και σε πολλών blogger που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Κάναμε διαβήματα και στις Βρυξέλλες και στην ε, Τεχεράνη ε, όποτε αυτό χρειάστηκε και έχουμε υιοθετήσει κυρώσεις εις βάρος 61 ε, ατόμων όσον αφορά την καταστολή στο Ιράν και συνεχίζουμε να το εξετάζουμε. Και τέλος μία λέξη για τον Νότιο Σουδάν γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία παρακολουθούμε στενά και για την οποία φοβούμαστε όσον αφορά την επιδείνωσή της. Όπως ξέρετε έχουμε μια συνολική προσέγγιση και στα δύο Σουδάν. Στόχος μας είναι δύο χώρες οι οποίες θα συνεπάρχουν ειρηνικά. Φαίνεται πως υπάρχει κάποια ε, κινητικότητα συνομιλίες βορρά-νότου και βεβαίως ε, είχα και μια επικοινωνία με τον ε, πρόεδρο Μπέκη της και χαιρετίζω τις ε, προσπάθειές του για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η συμφωνία συμφέρουν και τις δύο χώρες και στηρίζουμε τον πρόεδρο στις ε, προσπάθειές του. Επίσης χάρηκα για το ότι ο πρόεδρος όπως αφήνισε πως το Νότιο Σουδάν θέλει να ενταχθεί στην ε, Συμφωνία Κοτονού και μου το επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί που τον συνάντησα. Ελπίζω λοιπόν κύριε πρόεδρε να σα έδωσα μια ιδέα για πολλά από τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά βεβαίω ακόμα, οπότε θα σταματήσω εδώ πέρα, εάν μου επιτρέπετε, και θα σας παραδώσω το λόγο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντιπρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση, έχουμε πολλούς ομιλητές. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές να περιοριστούν σε δύο λεπτά ο καθένας και μετά έχουμε δύο ακόμη γύρους και εκεί οι ομιλητές θα μιλήσουν ένα λεπτό ο καθένας ε, για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Αλαφράνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε παρονιάστον. και να τα εκατοστήσετε. Ε, δεν ξέρω βεβαίω αν θέλετε πραγματικά να είστε εδώ πέρα. Θα προτιμούσατε να είστε κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει καλωσορίζω τις ε, δηλώσεις σας ε, για τις χθεσινές σας δηλώσεις για την επίθεση στην Τουλούζ. Πράγματι από ό,τι φαίνεται παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσει σας. Ε, η σημερινή διευκρίνηση πράγματι ξεκαθαρίζεται πραγματός όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Να ρωτήσω δύο πράγματα σήμερα. Συναντηθήκαμε με τον Παλαιστίνο Υπουργό Εξωτερικών που εξέφρασε την απογοητευσή του για την οικονομική κατάσταση τη... της Παλαιστίνης γιατί έχει περάσει η Παλαιστίνη σε δεύτερη μοίρα πίσω από την Αραβική Άνοιξη, τις Αμερικανικές και τις Ισραηλινές εκλογές και ανέφερε μια επιστολή προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό με στόχο να εκφράσει το ότι έχει ουσιαστικά πεθάνει η ειρηνευτική διαδικασία. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα. Τώρα όσον αφορά τη Ρησία. Οι Ρώσοι αντί να μετακινηθούν ε, θεωρούν πως ο νόμος πρόεδρος είναι ο πρόεδρος Ασάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα σχέδιο σε συνεργασία με τον Κόφι Ανάν, τον πρώην πρόεδρο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Θεωρείται πως μπορούμε να μειώσουμε τους θανάτους στη, στη Συρία. Τέλος, ο Βρετανό Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ ε, έκανε μια κοινή δήλωση με τον πρόεδρο τον Ομπάμα λέγοντας πως ε, το περιθώριο στενεύει συνεχώ για ειρηνικές διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το Ιράν. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Λέδη Άστον, και καλωσορίζω την ανακοίνωσή σας ότι θα υπάρξει και εκπρόσωπος θα διοριστεί είναι σημαντικό. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί στατηγικά. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα είναι απλώς λόγια. Σημαντικότατα αυτό τώρα που βλέπουμε τις δυνατότητες της εξωτερικής πολιτικής που πειράζεται αρνητικά από την οικονομική κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη εστίασης. Χρειαζόμαστε να ηγηθείτε, να μην φυστείτε προσπαθειών να πιέσετε τα κράτη-μέλη να μην είστε ντροπαλοί. Ερώτηση. Ιράν. Εκτιμούν τι προσπάθειε που καταβάλλεται να ξαναέρθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι έχει όμω ε, να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι απειλέ κατά τον ΗΠΑ και το Ισραήλ και τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ιρανικό λαό όσον αφορά τι κυρώσει που δεν έχουν σαν στόχο τον Ιρανικό λαό Στη Ρωσία ο Βίσμαρκ είπε κάποτε ότι η Ρωσία ποτέ δεν είναι τόσο ισχυρή ούτε τόσο αδύναμη όσο φαίνεται. Γίνονται αλλαγέ εκεί παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν ε, ξαναπαίρνει τη θέση του Τσάρου, ε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξακολουθεί ε, να, παρα... να οδηγείται στη σχέση με τη Ρωσία από οικονομικά συμφέροντα κάποιων χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, η Λιβύη. Ε, γίνεται, κάνετε πολύ σημαντική δουλειά ότι άνοιξε το γραφείο στην Βεγγάζη. Και υπάρχει και ιδέα για κοινό προξενείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βεγγάζη. Θα είναι πολύ σημαντικό για το λαό εκεί. Ελπίζω να ηγηθείτε αυτέ τι προσπάθειε και θέλουμε να υπάρχει και μόνιμο πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ενώση στην Τρίπολη για να μπορέσει να μιλεί με του Λίβιου διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα όσον αφορά το δυναμικό ανοικοδόμηση. Τώρα είναι η στιγμή σωστή. Θα γίνουν εκλογέ τον Ιούνιο. Πρέπει να γίνουν τα πάντα. Υποστήριξη τη προετοιμασία των εκλογών ε, και γενικά έχουμε αναλάβει θέματα όπως ασφάλεια των συνόρων μέσα της, ε, μεσικά μέσα ενημέρωσης, κοινωνία των πολιτών κλπ. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες. Ελπίζουμε όλη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα να μην χαθεί αν δεν συνεχίσουν οι προσπάθειες. Ευχαριστώ κυρία Νίτ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βαρώνει. Καταρχάς χρόνια πολλά. Δεύτερον, ήμουν παρούσα χθε στην ε, διάσκεψη ε, και άκουσα την ομιλία σας και επιβεβαιώνω ότι πράγματι δεν είπατε τίποτα όπως αυτά που θεωρεί ότι κατάλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών και δεν ήταν καθόλου καλά εμπνευσμένα τα σχόλιά του που απευθύνθηκαν εναντίον σας και τα απορρίπτω αυτά που είπε, διότι δεν είχαν καμία θέση. Θέλω να μιλήσω για την Αίγυπτο. Δείξαμε καλή βούληση, θελήσαμε να βοηθήσουμε την Αίγυπτο, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, υπήρξαν εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, άκρως ησυχητικές εξελίξεις, τα, στατοδικεία εξακολουθούν να δικάζουν πολίτες, καταδικάζονται με αυστηρότατες ποινές, κάποιοι θεωρώντας ότι έχουν προσβάλει τον στρατό και δεν ξέρω πώς θα γίνει η μετάβαση προς η μορφή δημοκρατίας. Άρα έχουμε πρόβλημα, δίλημα. Θέλουμε να υποστηρίζουμε τους Αιγυπτίους, τον Αιγυπτιακό λαό, αλλά δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι συμβαίνουν πράγματα και μερικά από αυτά είναι χειρότερα από αυτά που συνέβαιναν επί Μουμπάρακα. Όσον αφορά τη Συρία, έχουμε μια στάση παράξενη της Ρωσίας. Κατηγορείται ότι χορήγησε στρατιωτικό εξοπλισμό η Ρωσία στη χώρα και ταυτόχρονα όπως και ο Ερυθρός Σταυρός και η Ρωσία ζητά ανακοχή καθημερινή. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Ποια είναι η προσέγγιση σας όσον αφορά τη Ρωσία. Και τέλος, η γείτονα μου ζήτησε να ρωτήσω και το κάνω ευχαρίστω αν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το όραμά σας όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα γενέθλιά σας χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ που βρισκείστε αυτή τη μέρα σήμερα μαζί μας. Και το να έχουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνο. όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να σας ρωτήσω, στο μέλλον, ακόμα και αν υπάρχει ένας ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελπίζουμε εσείς να μιλάτε πολύ ανοιχτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε την τελευταία εβδομάδα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Καζακστάν, λίγες ώρες πριν υποβάλουμε το ψήφισμα, απελευθερώθηκε τελικά ένας κρατούμενος από τη φυλακή. Επομένως βλέπετε ότι όντως καταφέρνουμε να πετύχουμε αποτελέσματα όταν μιλάμε ανοιχτά για τη Συρία. Είπατε για την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρόσφατα, ένα ρωσικό πλοίο με όπλα, τα οποία πήγαιναν προς το καθεστώς Ασάντ, ουσιαστικά επιτρέπει και να περάσει ε, το διάβαστο πλοίο αυτού από τις κυπριακές αρχές. Επομένως, δεν άκουσα από εσά καμία επίκριση ως προς αυτό. Το ότι αφέθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ένα ρωσικό πλοίο να μεταφέρει όπλα προς το καθεστώς Ασάντ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν εσείς το γνωρίζετε αυτό, αν κάνετε κάποια δήλωση σχετικά με αυτό. Νομίζω θα πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά γιατί κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Όσον αφορά τώρα τα Βαλκάνια διάλογο ανάμεσα στο Κωσυφοπαίδιο και τη Σερβία. Ο διάλογο αυτό καταλήγει επιτέλου σε κάποια αποτελέσματα, σημειώνεται μια κάποια πρόοδο. Ωστόσο, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και τον κύριο Κούπερ για ό,τι έχει γίνει. Έχει σημειωθεί πρόοδο, αλλά δεν αρκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουν και τα δύο μέρη μετά τι σερβικέ εκλογέ του τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε ακόμα αρκετά ενωμένοι. Έχουμε όλη αυτή την πολιτική υποστήριξη και παρόλα αυτά υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη τα οποία δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου τέσσερα χρόνια μετά την δήλωση. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποβάλλετε κι εσείς την απαραίτητη πίεση προκειμένου οι χώρες αυτές τελικά να αναγνωρίσουν το κοσφοπέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα πω πω ε, κλείνει ο κατάλογο των ομιλητών. Δεν ξέρω ακόμα και αυτοί που έχουν εγγραφεί αν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι, εδώ είμαι και σβήνει το μικρόφωνο του κύριου Τάνοκ. Άκουσα τα σχόλια στον Ισραηλινό τύπο, είμαι φίλος του Ισραήλ και μόνο το μικρόφωνο του κύριου Τάνοκ έχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω πως ε, πράγματι υπήρχε κάποια παρεξήγηση. Hello, is that working now? Uh, sorry, I just... Δουλεύει. Ε, πράγματι υπήρξε κάποια παρεξήγηση των όσων είπατε. I have to keep my finger here, Ε, μα πρέπει να, το, να κρατάω το κουμπί πατημένο. Hello, yes, I don't know... Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τα όσα είπα, ε, αλλά υπήρχε πράγματι παρεξήγηση των όσων είπατε και εγώ βεβαίως θα ήθελα να προσθέσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δολοφοληθέντων των μαθητών και των στρατιωτών στη Γαλλία. Ελπίζω ο δολοφόνος αυτός κατά να ε, αντιμετωπίσει σύντομα τη δικαιοσύνη. Τώρα για τα σημερινά θα συμφωνήσω με την κυρία Νέιτς για το ότι η Αραβική Άνοιξη γίνεται αραβικός χειμώνας σε κάποια σημεία, ειδικά η εκλογή κάποιων σκληρών στην Αίγυπτο και η πίεση που ασκείται στις κοινότητες των κοπτών. Πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κοινότητες οι οποίες κινδυνεύουν εάν επαληθευτούν οι φόβοι τους και έχουμε ένα σύνταγμα βασισμένο στη Σαρία. Επίσης, στη Μέση Ανατολή έχουμε την δέκατη επέτειο της Αραβικής Πρωτοβουλίας για την Ειρήνη. Θεωρείται πως θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει αφορμή να ξαναξεκινήσει ένας λογικός διάλογος και να επανέλθουν όλα τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί πρέπει να καθησυχάσουμε του φόβου του Ισραήλ πω τώρα είναι περικυκλωμένο από ασταθή και εχθρικά καθεστώτα. Τώρα, για να επανέλθουμε λίγο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα τη συνεχιζόμενη φυλάκιση τη κυρία Τιμοσέγκο και ηγετών τη αντιπολίτευση, μεταξύ των οποίων και οι υπουργοί που κατά την άποψή μου υφίστανται επιλεκτική αντιμετώπιση από το καθεστώς του κυρίου Γιαννουκόβιτς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απελευθερωθεί η κυρία Τιμοσέγκο και για να επανέλθω στην πόλη μου, το Λονδίνο και την διάσκεψη περί Σομαλίας πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια ακρόαση με τον διοικητή της ε, Αταλάντα, τον ε, κύριο Ρόντο και θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τις ε, ερχόμενες ε, εβδομάδες για να βρούμε μια ε, λύση για, μια, για ένα σύνταγμα της Σομαλίας. Εγώ είμαι υπέρ της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης, δεν ξέρω η κυρία και αν έχει τα ίδια συναισθήματα όπως για το κοσφοπέδιο, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει μία συνεπή στάση εδώ πέρα. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας για την διάσκεψη αυτή και τέλος για την υπηρεσία σας. Α, τελείωσε ο χρόνο μου. Ε, με υπολογίσατε ότι δεν μιλούσα πριν με το μικρόφωνο. Καλώς ορίζω. Το ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα κάνετε κάποιον έλεγχο για το μέγεθος των ε, διμερών πρεσβειών των κρατών μελών για να μειωθεί το κόστος λόγω της ε, προσθέμενης αξίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για να μας διαβεβαιώσετε και μας που έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Σας ευχαριστώ, κυρία Ε, Ευχαριστώ. Ναι, δεν το άκουσα αμέσω. Ευχαριστώ που έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα για τη Λιβύη. Κυρία, στον ε, πολλές οργανώσεις όπως η Human Rights Watch για Χωρίς σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός ε, αναφέρουν εδώ και μήνες βασανιστήρια αφαιρέτως φυλακιστέντων. Ο δε... Η The Human Rights Watch μιλάει για διάφορα ένοπλα σώματα που κυκλοφορούν και στην Τρίπολη και αλλού και φυλακίζουν ανθρώπους, τους κάνουν ηλεκτροσόκ και τους βασανίζουν μέχρι θανάτου σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι γνωστά Επιπλέον, ο απεσταλμένος της νέας λιβικής κυβέρνησης στην πρώτη εμφάνιση ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επιτέθηκε ε, στους ομοφιλόφιλους και έτσι πλέον δεν μπορεί να γίνεται λόγος για οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μίλησε μάλιστα για το ότι αμφισβητείται η επιβίωση της ανθρωπότητας. Ε, θέλω να σας ρωτήσω, ε, αν γνωρίζετε αυτές τις ε, δηλώσεις και αν ε, τι προγραμματίζεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσουν τα βασανιστήρια και η παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως συνομιλητής και εταίρος και κυβέρνηση για τη Συρία. Πώς εκτιμάτε την αντιπολίτευση. Εγώ δεν έχω καταφέρει ε, να κάνω κάποια εκτίμηση. Στο ΝΑΤΟ και στην ΚΕΠΑ αναφέρεται πως ε, υπάρχει τώρα ένας νέος συνασπισμός της αντιπολίτευσης. Πώς βλέπετε αυτές τις διάφορες ομάδες και Ποιοι είναι οι συνομιλητές ε, της αντιπολίτευσης στην ε, Συρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να κρίνουμε την κατάσταση ε, την οποία πολλοί εκτιμούν ως εμφύλιο πόλεμο. Και τέλος, εκτιμάτε και εσείς πως υπάρχει εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, δεν ήσασταν εσείς οι μόνοι οι οποίοι μιλήσατε μισό λεπτό παραπάνω, αλλά από εδώ και μπρο θα είμαι πιο αυστηρός. Ο κύριος Μπέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, ε, χρόνια σας πολλά. Τώρα οι ερωτήσεις. Στο Βόρειο Ιράκ ε, υπήρξε μία εκδήλωση των κουρδικών φιλοδοξιών για αυτοδιάθεση και από ό,τι φαίνεται οι μειονότητες στην Τουρκία, Συρία, Ιράν και Ιράκ ε, ονειρεύονται ένα μεγάλο ε, Κουρδιστάν και δεν θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται εύκολη λύση σε αυτό το ζήτημα. Πώς το κρίνεται αυτό, θα μπορούσε να είναι πολιτικός δυναμίτης στη Μέση Ανατολή. Οπότε πώς βλέπετε τις ε, φιλοδοξίες περί Μεγάλου Κουρδιστάν. Δεύτερον, εκτιμώ τις προσπάθειές σας όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, στο Ιράν, αλλά θα είμαι πολύ περίεργος για την κατάσταση του Πάστορα Γιώζεφ Νανταρχάνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή το οποίο αυτή τη στιγμή η ζωή κινδυνεύει. Και τρίτη ερώτηση επίσης για το Ιράν. Ξέρετε πως ε, η κύρια ικανότητα των Ιρανών διαπραγματευτών είναι η αναβολή των διαπραγματεύσεων και όχι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή το ρολόι έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφη, αντίστροφα όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν. Και τέλος ε, η Συρία και η φρικτή αυτή η τραγωδία. Ένας ε, ιερέας έγραψε ε, αρχές αυτής της εβδομάδας πως είναι δραματική η κατάσταση των χριστιανών στη Χόμς και φοβάται ότι θα υπάρξει λουτρό αίματος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ασκήσετε κάποια πίεση για να αποφευχθεί μια τέτοια αντιπαράθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω διότι είναι ο πρώτος Γάλλος που παίρνω το λόγο σήμερα το απόγευμα. Να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε, για τη δήλωση που κάνετε την τραγωδία της Τουλούς. Αυτές οι διευκρινήσεις που κάνατε ήταν σημαντικότατες και αναμενόμενες. Το ερώτημά μου αφορά τρεις κρίσεις ή περιοχές κρίσης που μπορούν να θεωρηθούν ως περιφερειακές, αλλά εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναμειχθεί Σαχέλ, το κέρας Αφρικής και η Λιβύη. Είναι τρεις περιοχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ή την να αναπτύξει, θα έπρεπε να αναπτύξει την ε, προσέγγιση της στην παγκόσμια, τη σφαιρική. Εσείς ε, την εφαρμόζετε και την τροφοδοτείτε που είναι μια, ένα συν για την πολιτική μας της ασφάλειας, της άμυνας και της κοινή εξωτερική πολιτικής. Όμως έχω την εντύπωση ότι αυτή που επικρατεί από τις στατικές που εφαρμόζονται ή που θα έπρεπε να εφαρμοστούν σε αυτές τις ζώνες κρίσεων δεν είναι τόσο σφαιρική η προσέγγιση. Ε, έχουμε την πτυχή ανάπτυξη, την οικονομική πτυχή που λαμβάνονται υπόψη, αλλά η πτυχή της ασφάλειας δεν λαμβάνεται υπόψη χωρίς να μιλήσουμε για τη στρατιωτική πτυχή και την πτυχή της ε, ασφάλειας. Όμως αυτές οι περιοχές, Σομαλία πιο συγκεκριμένα, τις χώρες του Σαχέλ που πολεμούν την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα στη Λιβύη, όπου πήγαμε πρόσφατα, οι τοπικοί φορεί ζητούν κατεπήγοντος την συμπερίληψη της πτυχής της ασφάλειας στην πολιτική που απευθύνουμε προς αυτούς. Απευθύνω έκκληση προς εσάς, ούτω ώστε αυτή η σφαιρική παγκόσμια προσέγγιση να είναι σφαιρική γενική και να μην θυσιάζουμε την πτυχή ασφάλειας έναντι των άλλων πτυχών που είναι θεμητές και σημαντικές, αλλά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τις σε αυτή η πτυχή της ασφάλειας για να είναι χρήσιμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον θα αναφερθώ στα αποτελέσματα της διάσκεψης Γκίμνιχ, Χαιρετίζουμε το ότι θα υπάρξει ένα πακέτο, ένα ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα σχέδιο δράσης και μια πολιτική δήλωση. Αλλά δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένη με την πολιτική αυτή δήλωση. Αυτά τα οποία ακούσαμε είναι πως ε, απλά θα εγκριθεί ε, η ανακοίνωση του Συμβουλίου. Και μετά τη Λισαβόνα και τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, εμεί ε, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε μια κοινή δήλωση Κομισιών ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και σας παρακαλώ να καταβάλλετε λοιπόν κάθε σχετική προσπάθεια και να σκεφτείτε τι ε, άποψη έχετε για μια ομάδα εργασίας ε, από τα τρία θεσμικά όργανα που θα εργαστεί έτσι ώστε να έχουμε ένα τέτοιο έγγραφο. Και νομίζω θα έπρεπε να είναι έτοιμο τον Ιόνιο. Εάν δεν τα καταφέρουμε θα έχουμε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία αν ε, δηλαδή αναβληθεί για Δεκέμβρη κάπου εκεί. I think Νομίζω πως είναι καλή αυτή η ιδέα. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Λοιπόν, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ε, ευχές σας, για τα γενέθλιά μου και, ακόμη πιο σημαντικό, σας ευχαριστώ σε όσους με βοήθησαν να ξεκαθαρίσω τις χρησινές παρατηρήσεις. Ήταν ώρες δύσκολες για εμένα για το πώς ε, ε, παρερμηνεύτηκαν αυτά τα οποία είπα και σας ευχαριστώ που όσους ήσασταν εκεί και αν ε, κάποιος βεβαίως μπορεί να τα δηλώσει αυτά και δημοσίως θα ήμουν ευγνώμων για λόγους ευνόητους. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω στα ερωτήματα. Αν ξεχάσω κάτι, συγχωρήστε με. Κύριε Σαλαφράγκα, ξεκινήσατε με την συνάντηση με τον κύριο Μαλίκη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης ε, και την οικονομική κατάσταση και την επιστολή του Πρόεδρου Αμπάς. Πρώτα απ' όλα η Επιτροπή Ad Hoc ε, συνεδριάζει αύριο και εκεί πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την οικονομική κατάσταση. Εμείς ε, στηρίξαμε πάρα πολύ, όπως και πάρα πολλές χώρες, και το Ισραήλ, το έργο του Πρωθυπουργού Φαγιάντ για να οικοδομήσει τα θεσμικά όργανα ενός κράτους για να είναι σε θέση οικονομικά να προχωρήσουν και θα συνεχίσουμε να τους ε, στηρίζουμε. Έχουμε ήδη διαθέσει ε, κονδύλια για το μέλλον και ε, αυτό έχει τη, σημασία του. Αλλά βεβαίως δεν υποτιμώ την πρόκληση όπως είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Φαγιάντ χθες. Αντιλαμβάνομαι πως θα υπάρξει μια επιστολή του Προέδρου Αμπάς προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τον κύριο Νετανιάχου. Αντιλαμβάνομαι πως στόχο θα έχει να ξεκαθαρίσει την θέση του και να ζητήσει διευκρινήσεις. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρω και δεν ξέρω ακόμα πότε θα αποσταλεί αυτή η επιστολή. Αυτό το οποίο θα πω είναι πως ε, το ερώτημα το οποίο θέσατε για την όλη διαδικασία της Μέσης Ανατολής είναι πως συνεργαζόμαστε βεβαίως ε, στενά και με το κουαρτέτο ε, και αυτή τη βδομάδα θα συναντήσω τον απεσταλμένο αλλά και με τον Βασιλιά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιερδανίας, που εργάζονται ακούραστα για να ε, συναντηθούν άτυπα οι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές για να έχουν άμεσες ε, συνομιλίες. Οπότε υποστηρίζουμε την τοπική προσέγγιση, δίνουμε βάρος στο να έχουμε ε, ενορχιστρωμένες διαπραγματεύσεις και αυτό γίνεται στο περιφερειακό πλαίσιο που υφίσταται. Και σωστά βεβαίως αναφερθήκατε στη Συρία, στη Συρία και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί πέρα. Ε, ήμασταν ξεκάθαροι με τους Ρώσους, τους ζητήσαμε να επανεξετάσουν την ε, στάση τους για τα όπλα. Όχι μόνο γιατί τα όπλα τα χρησιμοποιεί το καθεστώς όπως ξέρουμε για να διαπράξει εγκλήματα, αλλά υπάρχει και κίνδυνος τα όπλα να πέσουν στα χέρια ποιος ξέρει πιανού και βεβαίως ε, αυτό από μόνο του δημιουργεί προκλήσεις. Δηλαδή ε, είναι ε, η παράδοση αυτή των όπλων οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση και επιμήκυνση της σύγκρουσης. Βεβαίως συνεχίζουμε τις επαφές με την Ρωσία και θα συνεχίσω να τονίζω αυτά τα πράγματα. Τώρα η συνεργασία με τη Ρωσία στην ανθρωπιστική πλευρά είναι επίσης σημαντική και βεβαίως γνωρίζετε τις προσπάθειες που γίνονται υπό την ηγεσία του Κόφι για να ε, έρθουμε σε επαφή με το Συριακό καθεστώς για τις ανθρωπιστικές ανάγκες και βεβαίως ε, είναι σε επαφή ο Κοφιανάν όπως και εμείς με τη Ρωσία για να προχωρήσουμε για τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Για το Ιράν, το παράθυρο της ευκαιρίας κλείνει. Αναφέρατε αυτά τα οποία δήλωσε, ε, δήλωσαν οι δύο ηγέτες στην Ουάσιγκτον. Ο ρόλος μου είναι σαφής. Εγώ υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να διευθύνω τις συνομιλίες ε, εξ ονόματος των ε3 Αυτή είναι η εντολή μου. Όλα τα άλλα δεν είναι δουλειά μου. Η δική μου δουλειά είναι να γίνουν αυτές οι συζητήσεις για να καταλήξουμε σε πραγματικά αποτελέσματα. Και τις συνομιλίες αυτές θα τις προσεγγίσω εάν γίνουν τις ε, ερχόμενες εβδομάδες, αν τις επιβεβαιώσουμε, με αυτό το πνεύμα θα τις ε, προσεγγίσω. Αναζητούμε μια λύση. Δεν πιστεύω πως θα γίνει με μια συζήτηση. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Κυρία Γκόμες, το να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για τις αποστολές. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να πιεστούν, να έρθουν σε επαφή με τις αποστολές που έχουμε και συναντιέμαι με πολλούς υπουργούς και με υπουργούς άμυνας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, ε, τις υφιστάμενες και οι νέες δεσμεύσεις βεβαίως να φροντίσουμε να ε, έχουν την σωστή στήριξη. Για το Ιράν, για τις ε, κυρώσεις ειδικά, είπα ειδικά για το Ιράν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κυρώσεις οι οποίες θα είναι σχεδιασμένες να πείσουν το Ιράν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μπορεί να έρθουν. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε σαφείς πως στόχος δεν είναι να πληγεί ο πληθυσμός του Ιράν και ο στόχος του να απαλλαγούμε από το πυρηνικό πρόγραμμα στηρίζει όλες μας φιλοδοξίες για έναν ασφαλέστερο κόσμο και αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για τη Ρωσία και τη στρατηγική προσέγγιση. Νομίζω πως όλοι τώρα με τον νέο πρόεδρο ε, που βεβαίως λογικό ήταν ε, είναι ο πρόεδρος Πούτιν ε, κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε υπάρχει εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό κάτι το οποίο επινόησε ο πρόεδρος Μπαρόζο στο... είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για μένα ως αντιπρόεδρο Συνεχίζουμε λοιπόν την δουλειά με τη Ρωσία όχι μόνο σε οικονομικά αλλά και σε πολιτικά ζητήματα και συνεχίζεται ε, η συνεργασία όπως πριν ως ένα βαθμό αλλά και διεθνώς είναι ένας ε, τομέας όπου όπως είπα οι στρατηγικές μας ε, συνεργασίες εφαρμόζονται και είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά το τι, μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Για τη δεν Βενγκάζη γνωρίζω πως ε, σας απασχολεί το ζήτημα και τώρα κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε ακριβώς και την περιοχή αυτή αλλά μην παρεξηγείτε εδώ πέρα τα πράγματα. Αυτά τα οποία έγιναν στην Τρίπολη δεν είχαν στόχο να απομακρυνθούμε από τη Βενγκάζη. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό άτομο που έκανε μεγάλη δουλειά και έδειξε τη σημασία αυτής της ε, πόλης αλλά δεν τίθεται ζήτημα πως ε, βεβαίως συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτή την περιοχή. Για τους λόγους που είπατε, η Τρίπολη είναι πολύ σημαντική. Κύριε Νέιτς, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για χτες. Η Αίγυπτος μας ανησυχεί ιδιαίτερα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα, ξέρετε, διαβάζω κάθε μέρα, κάθε λίγες μέρες ε, από τον επικεφαλή της αντιπροσωπείας τις εκθέσεις για το τι συμβαίνει ήμασταν σαφείς για την σημασία των ΜΚΟ και την σημασία του να υπάρχει η δυνατότητα της ελευθερίας του συνέρχεστε και είμαστε σαφείς γι' αυτό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα επίσης είμαστε υπέρ του να υπάρχει ένα σύνταγμα ισχυρό που θα προστατεύει το λαό και θα συνεργαστούμε με την Αίγυπτο καθώς προχωράει προς το μέλλον και πολιτικά και οικονομικά. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος ε, οικονομικά. Το ξέρουμε από τις επαφές μας, ε, εξετάζοντας το τι συμβαίνει στην οικονομία. Έχουν φοβερές προκλήσεις και γνωρίζουμε και εσείς και εγώ ε, από την αποστολή στην Τινησία όπου είχατε την καλοσύνη να έρθετε πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε όσον αφορά την οικονομική στήριξη της Αιγύπτου αλλά και την πολιτική στήριξη και να ασκήσουμε πίεση το ξεκαθαρίσαμε βεβαίως πως η χώρα είναι δική τους αλλά εμείς θα θέλαμε να δούμε δημοκρατία αυτή την οποία υποσχέθηκαν και στήριξη για την κοινωνία των πολιτών, για τις γυναίκες για να μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Ε, ρωτήσατε επίσης για την Κεντρική Ασία. Πήγα στην Αρμενία, στο Αζερβαϊτζάν και πραγματικά έχω δεσμευτεί για αυτές τις χώρες. Στην παρούσα στιγμή προσπαθώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε εκεί περιφερειακά. Προσπαθώ να δω αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική όπου υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπείες. Έχουμε πάντως καλές επαφές με το Κυργιστάν και με άλλες χώρες περιοχής και εκεί πέρα έχουμε διμερείς σχέσεις. Δεν σα λέω όμω ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω μια οριστική απόφαση, απάντηση με συγχωρείτε για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με την Κεντρική Ασία. Έχει ξεκινήσει πάντω η διαδικασία αυτή και θα επανέλθω για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική η περιφέρεια αυτή για μα. Κυρία Νουίντσεκ, ο ρόλος του ειδικού εκπροσώπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επηρεάζει καθόλου τον δικό μου το ρόλο. Πρόκειται απλώς για μία αναγνώριση ότι πρέπει να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα παγκοσμίω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν τόσες πολλές διεθνείς ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τόσες πολλές θεσμικές ευκαιρίες με τις οποίες πρέπει και εμείς να συνταχθούμε. Πώς δηλαδή μπορεί να εργαστεί η Ευρώπη στον κόσμο προκειμένου να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες στις οποίες εμείς πρεσβεύουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε και το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε και ελπίζω ότι και εσείς θα συνεργαστείτε με αυτόν τον ειδικό εκπρόσωπο και είμαι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Αναφέρθηκα ήδη στη Ρωσία και στη Ρησία, αναφέρθηκα επίση ήδη και στο ζήτημα των όπλων, ζήτημα το οποίο θίγω σε επαφέ που έχουμε με τη Ρωσία. Λέω ότι αυτό μα ανησυχεί πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα να ξεκαθαριστεί το ζήτημα αυτό. Σερβία και Κωσυφοπαίδιο. Αναφερόμουν συγκεκριμένα σε ένα ρωσικό πλοίο το οποίο πήγε στη Συρία με την άδεια της Κύπρου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επικρίνεται Είπατε για ένα ρωσικό πλοίο το οποίο πέρασε από την Κύπρο πηγαίνοντας στη Συρία. Το ζήτημα αυτό το έθιξαν κάποια κράτη-μέλη, αλλά ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δική τους εθνική αρμοδιότητα προς αυτό. Δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα άλλο πέρα από το ότι οι κυρώσει που έχουν αποφασιστεί θα πρέπει να ελοπιθούν πλήρως. Επομένως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λυπάμαι που δεν άκουσα αυτό που είπατε πριν από λίγο. Τώρα, όσον αφορά τη Σερβία και το Κοσφοπέδιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του διαλέγου, διαλόγου, με να επιτύχουμε κάτι το ιστορικό. Και ήδη αυτό που έχουμε επιτύχει είναι ιστορικό. Βέβαια, ο δρόμο τη υλοποίηση των συζητήσεων αυτών είναι ανώμαλο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να επιτύχει ο διάλογο αυτό. Πρέπει να καταβληθούν λοιπόν πολλέ προσπάθειε και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως και τις δύο πλευρές, γιατί η προσωπική δέσμευση και των δύο πρωθυπουργών ήταν πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να καταφέρουν να συνεχίσουμε τον διάλογο αυτό με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον πρωθυπουργό Τάτσιτς ιδίω είδαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε κάποιους τομείς όπως το εμπόριο που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Βασικός μου στόχος, και στο επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή, είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί η σχέση που έχουμε με το κοσφοπέδιο, θα ενισχυθεί η σχέση αυτή και το μέλλον του ουσιαστικά βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς αυτό νομίζω ότι συμφωνούν και τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ε, ολοκλήρωση των συζητήσεων στην, ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μάλλον συζητήσει οι οποίε ολοκληρώθηκαν χωρί κανένα πρόβλημα. Οι συζητήσει αυτέ φέρνουν το κοσμοπέδιο πολύ πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ε, μπορούν να επωφεληθούν πάρα πολύ από αυτό. Υπάρχουν κάποιε μονομένε χώρε οι οποίε για δικού του λόγου δεν αναγνώρισαν το κοσμοπέδιο, αλλά αυτή είναι δική του λόγοι. Κύριε Τάνεκ, ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε για τι ε, διευκρινήσεις αυτές όσον αφορά τη δήλωσή μου. Ξέρετε πώς εκφράζομαι και τι ήθελα να πω. Τώρα, κοινότητα των κοπτών. Το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει πολύ και στα πλαίσια της συνδιάσκεψης Γίμνιχ. Με αυτό άλλωστε ξεκίνησαν οι συζητήσεις που είχαμε όσον αφορά την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία θρησκευτική πίστης. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράστηκε επ' αυτού και αυτό φαίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εστάλησαν πολύ ισχυρά μηνύματα όσον αφορά την ελευθερία της πίστης, την εξιθρησκεία, τη συμμετοχή όλων των πολιτών, το να μπορούν να συνεπάρχουν συμφιλειωμένα πολλές θρησκευτικέ κοινότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διμερείς διάλογοι με επιμέρους χώρες όπου η κατάσταση είναι δύσκολη. Επίσης, ξέρετε ότι έχουν περάσει πια πάρα πολλά χρόνια στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την Αραβική Άνοιξη. Περιμένουμε λοιπόν να δούνε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα ήθελα να δω και πώς θα τοποθετηθούν όλες οι αραβικές χώρες, όχι μόνο αυτές οι οποίες έχουν κινητοποιηθεί Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε ένα απολογισμό του παρελθόντος και να δούμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε πολύ πιο απτά αποτελέσματα να αποφασίσουν και τα εμπλεκόμενα μέρη για το πώς θέλουν να προχωρήσουν. Με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανίας συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στην Πράγα, τον κύριο Κουσέγκο, και μιλήσαμε για την ανατολική εταιρική σχέση. Και σε κάθε πάντως ευκαιρία αναφερόμαστε στα ίδια ζητήματα. Η Γιούλια Τιμοσέγκο, αλλά όχι μόνο η Γιούλια Τιμοσέγκο, θα πρέπει να έχει μια δίκαιη δικαστική μεταχείριση και ανησυχούμε πάρα πολύ για την υφιστάμενη κατάστασή της. Οι συζητήσεις βέβαια αυτές συνεχίζονται συνεχώς και θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά την ε, Ουκρανία, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ήδη μια συμφωνία σύνδεσης έτοιμη. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ισχυρή σχέση. Πρέπει όμως και αυτοί να κινηθούν από τη δική τους την πλευρά και ξέρουν από πολιτικής πλευράς τι πρέπει να γίνει. Αναφερθήκατε επίσης στη Σομαλία και για τις συναντήσεις που είχατε με την επικεφαλής αποστολής Αταλάντα και τον ειδικό εκπρόσωπο. Είναι πολύ καλή η ομάδα αυτή και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά για να παρακολουθήσουμε όχι μόνο αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο Λονδίνο, αλλά και όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία χρόνια. Γίνεται τώρα μία συνάντηση ανάμεσα στους ε, γενικούς ε, γραμματείς κρατών μελών με τον κύριο για να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί καλύτερα η συνεργασία. Δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Προσπαθούμε, για παράδειγμα, να δούμε ποια είναι η ποιότητα των υφιστάμενων επιτόπου υποδομών. Ενδεχομένω να μπορούμε να κάνουμε κάποια περισσότερα πράγματα με ορισμένε χώρε. Το ίδιο είχε γίνει και με το Σουδάν, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία συνεργάζονταν από κοινού. Αναφερόμαστε λοιπόν στην ποιότητα των υποδομών και, να δούμε, και προσπαθούμε επίση να δούμε τι συνέργειε, βελτιωμένε συνέργειε μπορούμε να πετύχουμε επιτόπου. κυρία Λέσινγκ. Για τη Λιβύη είπα μερικά πράγματα. Το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο είναι ακριβώ αυτό που αναφέρει και η ονομασία του Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο και πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και ξέρετε ότι συνομιλούμε μαζί του να βρούμε λύσει, Υπάρχουν πραγματικέ δυσκολίε και ανησυχώ πάρα πολύ όπω και εσεί για την όλη κατάσταση σε κάποια τμήματα τη Λιβύη. Για τη Συρία αναφέρθηκα στην αντιπολίτευση και τις δυνάμεις της. Δεν θέλω τώρα να περιγράψω με ονόματα την κατάσταση. Θέλουμε να έρθω σε επαφή με όλες τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια προσέγγιση η οποία συμπεριλαμβάνει τους πάντες και ακολουθεί μια λογική προσφυγή. Πορεία. Κύριε Μπέλντερ, για το Βόρειο Ιράκ, δεν είμαι σίγουρο ότι μπορώ να περιγράψω τα θέματα συνομιλούμε με το Ιράκ. Το μεγαλύτερο θέμα πρόσφατα ήταν το στατόπεδά Άσραφ. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Ιράκ πάνω σε όλα τα ζητήματα και στο βορρά υπάρχουν προβλήματα γιατί αφορούν και την ενέργεια. Οπότε έχουμε ένα σύνολο ερωτηματικών εδώ για το Ιράν νομίζω ότι κολλησιεργούν οι Ιρανοί. Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί τους επί τη βάση της επιστολής του δόκτωρα Τζαλίλη, βάση της απαντήσεως που μου απέστειλε, πιστεύω ότι ίσως υπάρχει δυνατότητα συνομιλίας. Θα πρέπει να καταλάβετε όμως ότι ε, έχουμε ένα στόχο στις συνομιλίες και θα είναι σημαντικότατο αυτό να γίνει τάχιστα ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένας πραγματικός σκοπός στις συνομιλίες και αυτό για μένα θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας μπορούμε να ξεκινήσουμε με σεβασμό εναντί του Ιράν αλλά και σαφώς πρέπει να δηλώσουμε ότι θέλουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να δούμε πρόοδο. Κύριε Ντονζάν, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Αναφερθήκατε στη Λιβύη, το κέρας της ε, Αφρικής και το Σαχέλ, ναι, πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα από ό,τι μέχρι τώρα σε αφορά τι στρατηγικέ που θέλουμε να εφαρμόσουμε για το Σαχέλ. Έχουμε καλή στρατηγική, πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή τη. Για το κέρα Αφρική έχουμε μια ολιστική ισχυρή προσέγγιση, θα πρέπει να λειτουργήσει κάθε κομμάτι αποτελεσματικά για τη Λιβύη. Μαζί με τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα θέματα που μας απασχολούν. Συμφωνώ μαζί σας. Η κυρία Λοκλίμπε, πολιτική δήλωση. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να συμμετάσχω με τέτοια προσέγγιση. Δεν θέλω όμως να περάσει ένα εξάμεινο με συζητήσεις για κάποιες λέξεις. Το ξέρετε αυτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι ζωντανό. Είναι κάτι που αφορά αυτά που κάνουμε. Αν μπορέσουμε να βρούμε λοιπόν μια διέξοδο θα ήμουν ευγνώμων. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα τηρήσουμε το ένα λεπτό. Παρακαλώ να το τηρήσετε. Πρώτα απ' όλα κυρία Μούνιθ. Ευχαριστώ, Λέδη Άστον, που ήρθατε στη συνεδρίαση. Τώρα, επανερχόμενοι στη Μέση Ανατολή, έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς εφαρμόζεται αυτή η αρχή του περισσότερα για περισσότερα στο Ισραήλ, more for more. Θα ζητηθεί μια συμφωνία, να υπάρξει συμφωνία με το Ισραήλ για φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτά που αναφέρουν λοιπόν από την αντιπροσωπεία μας στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, μας λέγουν οι αντιπρόσωποι μας ότι γίνονται κατεδαφίσεις και νέοι επικισμοί. Οπότε οι θέσει του Ισραήλ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, είναι μια θέση παράλυσης θα έλεγα. Στην παρούσα κρίση υπάρχει το πρόβλημα και το εμπορίο όπλων. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι πίσω σε δεύτερη θέση μετά τη ΣΥΠΑ όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων. Η Γερμανία αύξησε τις πωλήσει όπλων προς τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Και κάποιες αραβικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ ότι ε, εξοπλίζει τρομοκρατικές ε, ομάδες. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η υποψή σας από αυτού, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ήπατη εκπρόσωπε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά σας να είστε εδώ. Δύο ερωτήσεις έχω. Χαιρετήσατε την εκλογή νέου Προέδρου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας μετά από μακροχρόνια κρίση και είπατε ότι σε αυτή τη δήλωση ότι αυτή ήταν η λύση της κρίσης στην υπερνηστερία. Περιμένετε και ας φωτοβουλίζει το θέμα. Κάνατε πρόσφατα μία επίσκεψη μετά στη Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία. Σαν εισηγητής για την Ισλανδία, με ενδιαφέρει να γνωρίζω την προσέγγισή σας για το θέμα της Αρκτικής. Και αν αναφέρθηκε η Ισλανδία στις συζητήσεις σας κατά το ταξίδι σας αυτό. Ευχαριστώ πύρος για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημά μου είναι απλούστατο. Λόγω της κρίσεως. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Λόγω της κρίσεως, θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη είναι πιο συνεργάσιμα ή λιγότερο όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση που αφορά την... αυτά που υπόθηκαν για τις κυρώσεις σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ένα σαφές παράδειγμα τη δημοκρατία της Λευκορωσίας. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα οι κυρώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε όλες αυτές οι παραβιάσεις που υπάρχουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως να σταματήσουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να σταματήσουν. Και κάτι άλλο που σχετίζεται με τη Λευκορωσία. Ελάχιστες προδιαγραφές που παραβιάστηκαν όσον αφορά τη θανατική ποινή και ότι οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να θάψουν τους νεκρούς του. Όσον αφορά αυτό το θέμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχετε να πείτε. Η κυρία Όγκολαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Μαρονιάστον. Το δικό μου το ερώτημα αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας για μια πιο συνεκτική πολιτική της Ένωσης όσον αφορά την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Εμείς ε, εκπλαγήκαμε από το θερμό χαιρετισμό σας για την εκλογή του κυρίου Πούτιν τη στιγμή που ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, ήταν πιο συγκρατημένος ή και επικριτικός και αργότερα το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ε, ένα ξεκάθαρο ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο λέγοντας πως δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες αυτές οι εκλογές. Οπότε θα ήθελα ε, να δω τη δική σας την άποψη ε, για μια πιο συνεκτική πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Κυρία Κρόνμπερκ. Έφυγε. Και ο Σκάμπελ Μπάνμαν. Βαρώνη. Να ρωτήσω την θέση σας για τα νησιά Φόλκλαντ. Είναι όλο και πιο επιθετική η Αργεντινή και πλησιάζουμε την 30η επέτειο της εισβολής. Κλασική συνταγή βεβαίως για να απομακρύνει την προσοχή από τον πληθωρισμό που είναι 20% επί Κίρχνερ. Έχουν περάσει αλληλευτικά τους ε, σκάφη στα ε, βρετανικά ύδατα, εμποδίζονται οι πτήσεις, ε, αλλά βεβαίως ε, τα αιτήματά τους ήταν ούτως ή άλλως φεδρά. Το 1592 ο Σερ Τζον Ντέιβις κατέκτησε αυτά τα κατοίκητα νησιά, δηλαδή πριν να υπάρξει καν η Αργεντινή. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε εμπορικές κυρώσεις, π.χ. αναστολή των εμπορικών συμφωνιών, ειδικά για το βόλιο κρέας και των διαπραγματεύσεων για ελεύθερο εμπόριο με τις χώρες Μερκοσούρ που υποστηρίζουν την Αργεντινή. Τονίστε επίσης στην πρόεδρο Κίρχινερ ε, πως δεν είναι σωστές αυτές οι δηλώσει. Ο πρόεδρος λέει δεν μπορώ εγώ να υποστηρίξω κυρώσει κατά του αργεντινικού βοήου κρέατος. Ε, η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μασπέλντερ για την κατάσταση των χριστιανών στο Ιράκ και των ε, ασυρίων που αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα το δεύτερο μου ερώτημα. Είπατε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά τα οποία ενώνουν όλες τις πτυχές της ε, πολιτικής σας. Σας ευχαριστώ για τις προσωπικές σας προσπάθειες ε, για το Αφγανιστάν ε, όταν είχαμε εκεί πέρα μία ενημέρωση για τις γυναίκες και τις γυναικείες φυλακές. Τώρα, Αναφέρατε ένα σχέδιο δράσης, έναν ειδικό απεσταλμένο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει βεβαίως ε, μία διαφορά μεταξύ ε, βεβαίως ε, των αποστολών όπου ο πρέσβης πρέπει να διατηρεί κάποιες καλές σχέσεις και των προσπαθειών που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία στον δύο χρόνια τώρα κάνετε αυτή τη δουλειά και πηγαίνετε ε, από τη μία άκρη της Ιφιλίου στην άκρη. Και δεν φτάνει ποτέ σε κανέναν. Ε, μόλις φτάσετε στο ένα σημείο πρέπει να σηκωθείτε να φύγετε για να πάτε σε ένα άλλο. Και το ερώτημα είναι, Εάν είναι αυτός ο σωστός τρόπος, όταν βλέπω ε, πως έχετε ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου και το τι έχει γίνει με την ε, Συρία το ζήτημα είναι το εάν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να λειτουργεί ως ένας κανονικός υπουργό εξωτερικών ή εάν θα πρέπει να ασχολείται με τον συντονισμό της πολιτικής ε, και το τι κάνει ο κύριος Ντεχούχτ και ο κύριος Πίμπαλξ. Να δείτε δηλαδή συντονισμό της πολιτικής της εμπορικής και της αναπτυξιακής. Κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι έχει πάει σε πάρα πολλές χώρες η κυρία Άστον. Επομένως, όσον αφορά την Αργεντινή και την Βραζιλία, πιο συγκεκριμένα, πώς έχουν τα πράγματα ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρ. Κατά την άποψή σας και μετά τις εξελίξεις που είχαμε την τελευταία εβδομάδα, και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν περισσότερο σε πραγματές αυτές πριν το καλοκαίρι. Θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πριν την σύνοδο που θα γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής τον Ιανουάριο. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Συγγνώμη, σκεφτόμουν τελευταία ερώτηση και δεν πρόσεχα. Σκεφτόμουν απλώς τελευταία ερώτηση. Σας ζητώ συγγνώμη. Κυρία Γκούνες, εσείς αναφερθήκατε με την πρωτοβουλία More for More, το Ισραήλ και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Γίνανε απλώς κάποιες συζητήσεις που ξεκινήσανε νομίζω το 2005 για το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ. Υπάρχει μια νομική βάση, εντάσσεται στην Συμφωνία Σύνδεσης και θα διαπραγματευτούμε με τον ίδιο τρόπο και με άλλες χώρες στο μέλλον. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μην παρερμηνεύουμε την συμφωνία αυτή. Και όσον αφορά τους επικισμούς, θα πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτούς να μπορούν να πάνε σε τόπους όπου θα μπορούσαν να, να ζήσουν μακροπρόθεσμα και ειρηνικά. Κύριε Σπράντο, εσείς αναφερθήκατε στην Μολδαβία και το πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση για την υπερνηστερία. Σε μια συνάντηση που έγινε στο Δουβλίνο 5 συν 2 το Φεβρουάριο συγκεκριμένα και θα έχουμε και μία ακόμα στην Βιέννη τον Απρίλιο τέτοια συνάντηση προσπαθούμε να αυξήσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν προκειμένου να βαθυθεί η συνεργασία με τους διεθνείς μας εταίρους και ιδίως με τη Ρωσία. Γιατί νομίζω ότι αν σημειωθεί πρόοδος θα σταλεί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και ελπίζω ότι με τον νέο πρόεδρο τώρα θα είμαστε σε θέση να δούμε να σημειώνεται μια πρόοδος. Επιτόπου προσπαθούμε να, να προχωρήσουμε κάποιες ιδέες οικοδόμησης εμπιστοσύνης προκειμένου να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών ιδίω. Ένα σημαντικότερο λοιπόν ρόλο επιτόπου και αυξημένη πίεση προκειμένου να συνεχιστεί η εργασία που έχει ξεκινήσει. Και πραγματικά θα ήθελα να ελπίζω και ελπί... ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αναφερθήκατε στην... στο ταξίδι που έκανα στην Αρκτική. Με έχει απασχολήσει η πολιτική Αρκτικής και θέλουμε να έχουμε και εκεί πέρα ένα μόνιμο εκπρόσωπο και ξέρετε ότι η περιφέρεια αυτή παρουσιάζει πάρα πολλά συμφέροντα, όχι μόνο επειδή έχουμε κάποια κράτη-μέλη που ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολύ σημαντικά συμφέροντα όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο, όσον αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα των περιοχών αυτών. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζουμε τι πιστεύουν οι κάτοικοι της περιοχής για την περιφέρεια αυτή και έχω πάει πάρα πολύ βόρεια προκειμένου να μιλήσω ακόμα και με επιστήμονες Γάλλους και Γερμανούς οι οποίοι εργάζονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφόρων στη Βόρεια Σουηδία για παράδειγμα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η, ε, ε, η συνάντηση αυτή. Δεν κατάφερα να πάω στην Ισλανδία. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια ισχυρή και ξεκάθαρη πολιτική για το μέλλον γιατί η περιφέρεια αυτή θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο μέλλον. Ε, κύριος Πάσκου, αναφέρθηκε στα κράτη-μέλη. Ναι, τα κράτη-μέλη συνεργάζονται όπως μπορούν στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι συνεργάζονται περισσότερο τελικά, είναι πιο συνεργάσιμα. Να σας πω και για ποιο λόγο. Ανεξάρτητα από το οικονομικό κλίμα, τα κράτη-μέλη βλέπουν ότι υπάρχει μια πραγματική αξία στη μεταξύ του συνεργασία νομίζω ότι τάσσονται υπέρ του να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι επικεφαλής των συζητήσεων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οποίος χαράσει πολιτική, συνεργάζεται μαζί τους και στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας τους επιτρέπει να περάσουν με ένα πιο συνεπή τρόπο το μήνυμά τους. Σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούμε κυριαρχία από τα κράτη-μέλη, καταφέρνουμε απλώ να συνεργαστούμε καλύτερα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμα. Κύριε Πυρσπίκ, αναφερθήκατε στις κυρώσεις και ιδίως στη Λευκορωσία και για την ε, η κατάσταση που έχουμε εκεί και στο Γκίμιχα συζητήσαμε το ζήτημα αυτό της απομόνωσης και της δέσμευσης. Πολύ συχνά κινούμαστε ανάμεσα στα δύο. Μέσω των κυρώσεων προσπαθούμε να στείλουμε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό και οικονομικό μήνυμα για μια χώρα. Και με τη Λευκορωσία η στάση μας ήταν ξεκάθαρη και θα συνεχίσει να είναι ξεκάθαρη. Είμαστε όμως σαφείς και για το πολιτικό μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε. Τι πρέπει να κάνουν. Θα πρέπει να αποφαλακιστούν αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να επιστρέψουν οι οικογένειές τους θα πρέπει πραγματικά να ελοποιήσουν τα όσα θεωρητικά λένε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Και αυτό που τους λέμε είναι ότι αν τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, τις υποσχέσεις σας, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό το μήνυμα στέλνουμε και μέσω της Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω των κρατών μελών που μονομένα έχουν επαφές στη Λευκορωσία. Στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα αυτό, κάνουμε ό,τι κάνουμε γιατί θέλουμε να αλλάξετε. Και αν αλλάξετε είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη γραμμή αυτή, να ακολουθούμε αυτή την πολιτική. Κύριε Άτσαλαντ, αναφερθήκατε στην Ρωσία. Δεν είπα, δεν χαιρέτησα, κατέγραψα το γεγονός ότι ο κύριος Πούτιν είναι ο νέος πρόεδρος και η στάση μου ήταν απόλυτα στονισμένη με τον κύριο Σούλτς. Επίτηδες, γιατί ξέρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό και έπρεπε να σταλεί με τον σωστό τρόπο υπάρχει γενικότερη αποδοχή ότι ο κύριος Πούτιν είναι ο νέος πρόεδρος της Ρωσίας που είχε κλεγεί από το λαό. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα τα οποία και εσείς δηλαδή της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τη Ρωσία. Το σημαντικό είναι να καταγράψουμε τι έχει συμβεί και να προχωρήσουμε. Και κάνοντας κάτι τέτοιο, η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών της Ρωσίας μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο κύριος Κάμπελμπαν. Αναφερθήκατε στα Φόλκλαντ. Ξέρετε ότι πρόκειται για διμερές ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο αφορά κυρίαρχα το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πήγα στην Αργεντινή, πήγα στη Βραζιλία. Θα μιλήσω σε αυτό, γι' αυτό σε λίγο. Σε καμία περίπτωση θα μπορούσαν να αποφασιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορικοί περιορισμοί η Γενική Διεύθυνση μπορεί να είναι σε επαφή πάντως μαζί τους και σας έχουμε πει και στο παρελθόν ότι είναι πολύ σημαντικό η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να, να εργάζεται για το ζήτημα αυτό που είναι καθαρά εμπορικό και όχι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Χριστιανοί τώρα στο Ιράκ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως σας είπα πριν από λίγο, στα πλαίσια της Συνόδου Γκυμνίχα αναφερθήκαμε πάρα πολύ στην υποστήριξη των θρησκευτικών μειονοτήτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται και πόσο σημαντικές επίσης είναι οι κοινότητε των χριστιανών στο Ιράκ και στη Συρία. Γι' αυτό το λόγο στείλαμε και αυτό το μήνυμα της ενοποιημένης κοινωνίας, τη συμμετοχής όλων των πολιτών. Απευθυνόμαστε σε όλου του πολίτε. Όλοι πρέπει να έχουν ένα μέλλον στη Συρία, όλοι θα, μπορούν, όλοι θα πρέπει να μπορούν να εξασκούν την πίστη τους ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει εμείς συνεχώς να στέλνουμε. Πρόκειται για ένα πολύ θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πολύ σωστά το θίξατε κι εσείς. Κυρία Σαρτζεντίνη έφυγε, θα απαντήσω, δεν τη βλέπω, να απαντήσω στο ερώτημά της όσον αφορά την συνοχή πολιτικών, εμπόριο ανάπτυξη. Αύριο θα συνδυάσουν οι επίτροποι Ρέλεξ ε, υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βαρόσο και εγώ θα συνεργαστώ μαζί του για να φέρουμε αυτή την ε, επίσημα την συνοχή, την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και στα διάφορα γραφεία των Επιτρόπων δημιουργήσαμε σχέσεις για να συνεργαζόμαστε με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Έχω υπόψη μου ότι ήμουν επίτροπος και είμαι επίτροπος ε, και έχω σαφή ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, στο τέλος της θητείας μου, εκείνος που θα με αντικαταστήσει, ίσως να μην έχει αυτό το παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα θα πρέπει ε, το έργο του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριληφθεί και να παγιωθεί εντό Επιτροπή Εξωτερική Δράση, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αυτό το στόχο έχω θέσει φέτο. Ότι πρέπει αυτό να το προωθήσουμε. Μετά για Βραζιλία και Μερκοσούρ. Είναι θέμα εμπορικό. Δεν θα έλεγα ότι ανήκει σε αρμοδιότητέ μου. Είναι αρκετά αργή η πρόοδο. Πού πήγε, Α, τον έχασα. Πού ήταν ο κύριο Γιάννη. Ζητώ συγγνώμη κύριε Γιάννη, δεν ε, είδα το όνομά σα. Λοιπόν, αργή η πρόοδο των διαπραγματεύσεων έγιναν κάποιες διευκρινήσεις. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα επί διαφόρων θεμάτων. Αλλά υπάρχουν προβλήματα συντονισμού από πλευράς Μερκοσούρ. Θα το εξακριβώσω κατά πόσο είναι αληθές. Πριν το τέλος του έτους θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και θα γίνει και άλλη μια σύνοδο καλοκαίρι. Οπότε ελπίζω έτσι να απαντώ σε αυτά που με ρωτήσατε. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα στα γενέθλιά σας ήρθατε εδώ πέρα. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν πήραν τον λόγο. Αυτό οφείλεται σε αυτούς που μίλησαν παραπάνω. Δεν θα το επιτρέψω την επόμενη φορά για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να μιλήσουν. Για να είμαστε και δικαίοι. Θέλω να ευχαριστήσω και σας αγαπητή κυρία Βαρόνη για το ότι είπατε πως το μέσο εταιρικής σχέσης είναι ουσιαστικό μέσο εξωτερικής πολιτικής και θα κινηθείτε αναλόγως και επιτρέψτε μου αγαπητοί συνάδελφοι να σας παρακαλέσω ε, να σηκωθούμε εις μνήμη των θυμάτων της τουλούς για τα νεκρά παιδιά του σχολείου και τους τρεις ε, δολοφονημένους αλεξιωτιστές. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Λίγα τη συνεδρίαση.